Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, βελτίωση τη οικονομική διακυβέρνηση και του πλαισίου σταθερότητα τη Ένωση, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Και ο εισηγητή είναι ο Διόγκο Φέιο, έχει εκπονήσει ένα έγγραφο εργασίας. και Φέη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε το έγγραφό σας. Ευχαριστώ. Σε, σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψε, κυρία Πρόεδρε, και στα πλαίσια μιας έκθεσης, η οποία έχει σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση και τη ευρωπαϊκή σταθερότητα στην ΕΠΣ, ιδιαίτερα το χώρο του ευρώ, θέλω καταρχήν να υπενθυμίσω την προέλευση αυτής της έκθεσης. Μετά από μια οικονομική κρίση διεθνή την οποία έχουμε υποστεί όλοι, η οποία είχε επίπτωση και επιπτώσεις επί της Ευρώπης και η οποία μας οδήγησε να συμπεράνουμε πως η καλύτερη αντίδραση της ζώνης ευρώ ήταν να πάρει μερικά μέτρα. Αν και με αυτά τα μέτρα ήταν αργά και αν δεν είχαν τα ευκαιρία αποτελέσματα. Ωστόσο, ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτή την κρίση σαν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία που θα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε εις βάθος ένα σύνολο διαδικασιών. Αυτή η κρίση επίσης θα πρέπει να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε ορισμένους τομείς και να κάνουμε πρόοδους. Το Μάιο η Κομισιό έκανε μια ανακοίνωση η οποία πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια του Συμβουλίου υπό την προεδρία του Βαν Ρομπέι δημιουργήθηκε μια task force μια ομάδα κρούσης και το Κοινοβούλιο είπε ότι θα πρέπει να είναι παρόν και θα πρέπει να πάρει μια θέση η οποία θα είναι σταθερή, μόνιμη, ενεργή και νομίζω πως πραγματικά είναι, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες σε αυτά τα θέματα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Επίσης υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τίθενται και ερωτήματα σε, και ένα από αυτά είναι ποιος θα είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος θα είναι η καρδιά της αντίδρασης σε αυτή την προσπάθεια κατά πόσον θα πρέπει να είναι πιο φεντεραλιστική, ομόσπονδη δηλαδή ή κυβερνητική. Είναι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τα πουλαράζα το παρελθόν, ιδιαίτερα εφόσον εμφανίζονται πολλοί σε αυτό το κοινοβούλιο και αλλού οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις ωστόσο πρέπει να έχουμε μια θέση ενιαία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτό, αυτού και είναι δυνατό το κοινοβούλιο να παρουσιάσει το καλοκαίρι μια τέτοια θέση η οποία θα είναι ενιαία και μόνιμη Ποιε είναι οι προκλήσεις τώρα οι οποίες μας αναμένουν στα πλαίσια τη συνάντηση την οποία είχαμε με τον κύριο Τρισέ μια κάποια στιγμή αναφερθήκαμε και διερωτηθήκαμε τι είναι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ευρωπαϊκή οικονομική συγγνώμη διακυβέρνηση. Και από αυτό το σημείο μπορώ να σας υποσχεθώ πως αυτή η έκθεση δεν θα είναι ένα θεωρητικό πόνημα αλλά θα είναι μια έκθεση η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη, η οποία θα, το οποίο θα παρουσιάζει ορισμένες δράστης, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, δραστηριότητες οι οποίες και δράσεις μπορούν να αναπτυχθούν επί του θέματος αυτού και όταν μιλούμε για το βραχυπρόθεσμο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ότι είμαστε στα όρια της συνθήκης της Ένωσης Δηλαδή έχουμε μια πρώτη πρόκληση η οποία έχει σχέση με την νομοθεσία και με την παράγωγη νομοθεσία η οποία θα προκύψει από αυτό. Ιδιαίτερα επισημένοντας όλες εκείνες τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας και αναμένουμε. Η οικονομική διακυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθεί στο χώρο του ευρώ, στην ευρωζώνη, αυτό είναι το ερώτημα, ή αντιθέτως θα πρέπει να επικεντρωθεί στο σύνολο της ΕΕ των 27. Είναι αυτή η θέση την οποία εγώ υποστηρίζω. Θα πρέπει να συμμετάχουν και 27 με πτυχές οι οποίες θα είναι ειδικέ, οι οποίες θα πρέπει να άπτονται μόνο τη ζώνης, ευρώ. Άλλη πρόκληση είναι η θεσμή αυτή καθευτή. Ποια, ποιο θα είναι το θεσμικό κοινό όργανο το οποίο θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και φυσικά φρονώ πως θα πρέπει να είναι η Κομισιόν δεν νομίζω πως πραχυπρόθεσμα θα ήταν αναγκαίο να παρουσιάσουμε καινοτομίε θεσμικές. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα. Καθότι αυτό το οποίο μου φαίνεται πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να δράσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Πράγμα το οποίο μας οδηγεί τη συζήτηση την οποία ανοίγουμε αυτή τη στιγμή και η οποία θα ξεκινήσει στα πλαίσια αυτή την έκθεση, ποια θα είναι εκείνα τα μέτρα εμφάρισης που θα πρέπει να δοθούν σε σχέση με τα ελλείμματα και με το χρέος. Το ευρώ και το δημόσιο χρέος δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε που δεν είναι. Διότι πάντα υποστηρίξαμε και μιλήσαμε στα πλαίσια του ελλείμματος για το θέμα της σταθερότητας. Δυστυχώς, η δημόσιο δανεισμός παρελήφθη. Και είναι ένα μάθημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρουμε, να μάθουμε και μια ακόμη φορά να επανέλθουμε στη συζήτηση εκείνη η οποία άπτεται του ευρώ και σχέση ευρώ με δημόσιο χρέος και πού οφείλεται αυτό το χρέος και τι επίπτωση έχει επί της ε. Νομίζω λοιπόν η πρόκλησή μας είναι οι δομικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Μιλάμε για αυτές, μιλάμε επίσης για μια ανάγκη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και πάρα πολύ ειλικρινά σας λέω πως το σύμφωνο, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ασχολήθηκε πολύ με τη σταθερότητα αλλά ελάχιστα με την ανάπτυξη. Ξεχάσαμε και παραλείψαμε το θέμα ανάπτυξη το οποίο εκπροσωπεί τη μεγάλη πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η ΕΕ και την αντιμετωπίζει για το μέλλον. Θα πρέπει επίσης με ένα πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο να αξιοποιήσουμε και να δούμε ποιε θα είναι αυτέ οι αλλαγέ οι οποίε θα πρέπει να γίνουν σε αυτή την ανάπτυξη και βεβαίω θα μπορώ να σα μιλήσω καλύτερα για την Πορτογαλία, την οποία γνωρίζω καλύτερα. Ένα σύνολο μέτρων έχει ληφθεί αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, η τα οποία είναι μέτρα σαφή. υπάρχει αύξηση της φορολογίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ε, περικοπές όσον αφορά τις επιδοτήσεις τις κοινωνικές συγγνώμη, και φρονώ πως θα πρέπει να ξαναδούμε τα όρια τέτοιου είδους μέτρων τα οποία λαμβάνονται. Πού σταματάνε αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, μεγάλους στόχους, τους οποίους εμείς υποστηρίζουμε. Τέλος, η οικονομική διαχείριση θα πρέπει να μας επιτράψει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το ευρώ, το ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει όλο το πλαίσιο να ενισχυθεί αλλά και να τροποποιηθεί. Να τροποποιηθεί και να ενισχυθεί. Με τα εθνικά κοινοβούλια εμείς θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξουμε το ρόλο όσον αφορά τη διαφάνεια. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή θεσμικά όργανα με τα οποία μπορούμε να έχουμε Μάλλον έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσκολία να έχουμε την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ο λόγο τον οποίο πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση θα είναι ένα μεγάλο σήμα για ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία, προ τα άλλα θεσμικά όργανα και τα κοινοβούλια βεβαίω, καθώ επίση και την ανάγκη την οποία υπάρχει ότι θα πρέπει να είμαστε διαφανεί και δημόσιοι. Να υπάρχει δημοσιότητα δηλαδή, θα πρέπει να εξετάσουμε να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα εγγράψουμε στην έκθεση. Περαίνοντα λέγω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψει των υπολείπων συναδέλφων ευρωβουλευτών και έχω τη δυνατότητα να, είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με το σκιώδη εισηγητή ασπαζόμεθα όλη την ίδια άποψη και είναι πιθανό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσει μια θέση η οποία θα είναι ισχυρή, καινοτόμος, συνεκτική σε σχέση με αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Νομίζω πως είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και με τη βοήθεια όλων μας θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. νομίζω πως είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο θα ήθελα να ακούσω αυτή τη στιγμή τις παρατηρήσεις των συναδέλφων λέγοντας πάλι πως αυτή η κρίση είναι μια πρόκληση αλλά και μια δυνατότητα για την Ευρώπη να πάει μπροστά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει το ρόλο του στο μέτρο του δυνατού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω τώρα στους σκιώδους. Η Ελίζα είναι πρώτη σκιώδης της Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φέγιο διότι κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ανταλλαγής απόψεων ήδη παρουσίασε μια έκθεση, μια προέκθεση θα λέγαμε, ένα σχέδιο εκθέσεως και νομίζω πως η προθεσμία μεταξύ της παρουσίας αυτής της ανταλλαγής απόψεων και της παρουσίασης της πρώτης εκθέσεως είναι πολύ μικρή για μια έκθεση υψής της σημασίας. Ωστόσο θα ήθελα να πω πολύ σαφώς πως σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχουμε ενώπιόν μας μια σωστή βάση, μια βάση η οποία αποτελεί μια καλή έκθεση, αποτυπώνεται μια καλή έκθεση και πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Διότι προ στιγμή δεν, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη στιγμή, ούτω ώστε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα είναι πολύ πιο σταθερό για την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών και για την ΕΕ και να επιτρέπει μία, ένα συντονισμό και στο μέτρο του δυνατού να βάλουμε κάτι σε σε λειτουργία το οποίο θα είναι μια οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικότατο, ουσιώδη ρόλο καθότι βλέπουμε πως η βούληση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων είναι Βλέπουμε ποια είναι και αυτό είναι ο λόγο τον οποίο η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι μια συνενετική έκθεση και το υπογραμμίζω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Δεύτερη παρατήρηση είναι το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα ανοίγματο το οποίο υπάρχει και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλέ εκθέσει, πολλέ θέσει έχουν παρουσιαστεί εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε ενώπιον πολιτικών κομμάτων, ομάδων, τα οποία είναι διαφορετικά. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι το Κοινοβούλιο, λέμε όλοι, ότι θα πρέπει να έχει μια θέση αποφασιστική, σαφή. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε μια συνένεση. Και πιστεύω πως είναι πολύ πιο σημαντικό σήμερα να γίνει κάτι τέτοιο, λαμβανωμένη υπόψη παρούσα καταστάσεω. Όλα αυτά για να πω πω η έκθεση αυτή αφορά σε πολλά σημεία επί των οποίων εγώ προσωπικά και εκ πολιτικής μου ομάδος ε, θα πάρα πολύ μέτρα πρόληψης, μια εξισορρόπηση μεταξύ του δανεισμού και του ελλείμματος, στάθμισης των διαφόρων αυτών στοιχείων και εξισορρόπηση αυτών των σημείων και θα ήθελα να το ακόμη ότι θέλουμε να εξετάσουμε ορισμένα θέματα τα οποία είχαν μείνει σε δεύτερο πλάνο όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά στο μέτρο των μέτρων, των νόμων οι οποίοι ελήφθησαν. Είναι λοιπόν να καταλάβουμε ποια είναι η ανάπτυξη, είναι τα όρια, ποια είναι τα όρια, ποιος μπορούν, πώς μπορούν να αναπτυχθούν όλα αυτά τα πράγματα και αυτό το παραλαμβάνουμε πολλές φορές εδώ πέρα, χωρίς να ξέρουμε περί σου ομιλούμε πολύ συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τη διαφάνεια και την ασφάλεια, την ασφάλεια των στατιστικών στοιχείων και θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε ένα σύνολο οργάνων, μέτρων, τα οποία θα είναι πολύ σαφή και εγώ συμφωνώ με αυτά όλα. Φρονώ λοιπόν δεν θα πρέπει να χάσουμε πολύ χρόνο αναφερόμενος σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Θα μπορούσα εγώ να το κάνω σε μια συζήτηση την οποία θα έχω με τον εισηγητή και, και μέσα σε ένα πνεύμα το οποίο έχει υπογραμμιστεί στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής της εκθέσεως. θέλω ακόμη να επιμείνω και να πω πως στο σημείο 1 και 2 δεν βρίσκουμε κάποια οργάνωση των διαφόρων θεμάτων για να είναι αυτά τα θέματα πιο σαφή, καλύτερα οργανωμένα. Πιστεύω λοιπόν το σημείο 1 και 2 είναι αρκετά μεγάλα η σύσταση από την 3 μέχρι την 8 και νομίζω πως το στυλ του δεύτερου μέρους της έκθεσης συνάδει περισσότερο με, νομική εκείνη, με το νομικό εκείνο πλαίσιο και την νομική διαδικασία που υπάρχει και στη σύσταση 1 και 2 θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε για να γίνουμε πολύ πιο σαφείς να επεξηγήσουμε το ρόλο και τη θέληση να εξετάσουμε όλες αυτές, τα, όλες αυτές τις παραμέτρους οι οποίες δεν είναι σταθερές για τη μακροοικονομία και πιστεύω πως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο όχι να τα ελέγξουμε, να τα συνδυάσουμε με την πραγματική οικονομία, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέπει στην πράξη να παρακολουθήσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι αναπτύσσονται και υπάρχει μια άλλη διάσταση που είναι σημαντική και είναι η εξέλιξη των, της σύγκρισης της απόκλησης εντός της ΕΕ καθότι στα πλαίσια αυτών των ελλημάτων και του δανεισμού παριστάμεθα σε πιέσεις οι οποίες υπάρχουν ε, και οι οποίες προκύπτουν από την πραγματική οικονομία και οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη σε, σε σχέση με δείκτες οι οποίοι επηρεάζουν την οικονομία. Φρονώ λοιπόν πως είναι σημαντικό να γίνουμε πολύ πιο σαφείς, να υπάρχει μια ακόμη σαφέστερη διασύνδεση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται και αποφασίζεται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των ομάδων εργασίας μεταξύ του Task Force, του ΡΟΠΑΙ και στα πλαίσια της εκθέσεως όσον αφορά την κρίση με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα είναι συλλεκτικό και να ακουστεί. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο και αν υπάρχει μια υπερβολή λόγω της ελλείψης πληροφόρησης ε, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αντιπαραγωγικό και θα πρέπει να ορίσουμε τους στόχους, ποιους στόχους θέλουμε να φτάσουμε, να επιτύχουμε και να δούμε ποιες είναι τα, οι κυρώσεις ή τα άλλα μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρχουν. Πιστεύω λοιπόν πως η έκθεση αυτή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και θα είναι δυνατόν να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα συνένεση μεταξύ των βουλευτών και ευελπιστώ πως ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτή τη διαβούλευση και στις εργασίες οι οποίες γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σαρμόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα μιλήσω ισπανικά. γιατί και στα ισπανικά μιλήσαμε με τον Διάγκο Φέιο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Προσωπικά προσυπογράφω μέγα τμήμα της έκθεσης και δεν βλέπω να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για να την υιοθετήσει και η ομάδα μου σε μεγάλο βαθμό. Στο σημείο 5 γίνεται λόγος για δημοσιονομικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί μου λείπει κάτι. Δεν γίνεται αναφορά ε, σε μια ενιαία ευρωπαϊκή υπηρεσία σαν Υπουργείο Οικονομικών ή εφορία αργά ή γρήγορα. Θα πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Κάπου θα πρέπει να αρχίσει να μιλάμε για ένα εργαλείο που θα βελτιώσει την κοινή νομισματική πολιτική και είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την κοινή διακυβέρνηση και τη, της δίνει σάρκα και οστά. Είχε έρθει η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τις κρίσεις ευκαιρίες Θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε τις κρίσεις για να κάνει ποιοτικά άλματα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σήμερα δεν το βλέπω τόσο πολύ σαφές αυτό. Ολοκληρώνουμε το τριμερή διάλογο για το πακέτο της ε, χρηματοπιστωτικής εποπτείας και έχουμε το εξή δίλημα. Εάν το Κοινοβούλιο θα δεχτεί ή θα διατηρήσει τη θέση τη Ευρωπαϊκή ισχυρή εποπτείας ή απλώ εάν θα επαναπαυθούμε ή θα υποχωρήσουμε σε ένα συντονισμό των εθνικών ε, συστημάτων. Είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Χωσέ Μαρία Μαργκάγιο στην έκθεση που είχε κάνει το 2000 για την ανάγκη μιας κοινή ευρωπαϊκής ε, χρηματοπιστωτικής εποπτείας γιατί είναι ολοκληρωμένε πλέον οι χρηματαγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σήμερα όταν συζητούμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι πριν από 10 χρόνια ήδη το Κοινοβούλιο πρότεινε αυτό που χρειαζόταν η ευρωπαϊκή οικονομία για να αποφύγουμε χρηματοπιστωτικές κρίσεις του τύπου και της ένταση που ζούμε σήμερα. Αν δεν πούμε τίποτα λοιπόν, αν δεν αναφέρουμε καν αυτό το θέμα, εάν δεν μελετήσουμε λίγο αυτό το σύστημα, δεν λέω να είναι γενική εφορία, ένα φόρο να χειρίζεται, εν πάση περιπτώσει, και να ε, εκδίδει ευρωομόλογα μόνο για τα ευρωπαϊκά δημόσια έργα ή όχι να τρέχει να, να σώνει χώρες που δεν έκαναν ό,τι έπρεπε στο σύμφωνο σταθερότητα. Αλλιώ νομίζω χωλαίνει πάρα πολύ η έκθεση και το σύστημα ολόκληρο, αν δεν το αναφέρουμε καν. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε ε, Φέιο για την εξαιρετική σας εργασία και επειδή μας είπατε τη σκέψη σας για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε μια συνένεση γιατί βεβαίως ε, η αηφορία και η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ακούσαμε χθε τον κύριο Τρισέ, τόνισε την ανάγκη ενισχυμένης ε, δημοσιονομικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας. Ε, αν το είχαμε αυτό δεν θα ε, χρειαζόμασταν τέτοιου είδους έγγραφα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα-ένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την κατεύθυνση, για τον προσανατολισμό της έκθεσή σας και τη σύγκριση που κάνετε μεταξύ χωρών εντός και εκτός Ευρωζώνης. Είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση σε μεγάλο βαθμό και ειδικότερα ο, εμείς ε, που δεν ε, ε, συμμετέχουμε στο κοινό νόμισμα. Ευχαριστούμε πολύ για το σεβασμό των Εθνικών Κοινοβουλίων και της επικουρικότητας, γιατί νομίζουμε ότι και αυτό είναι σημαντικό. Χαιρετίζουμε τα βήματα για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χαίρομαι επίσης που αναφέρεται την, το να παραμείνουμε στην ε, ισχύουσα συνθήκη γιατί κάποια κράτη-μέλη μιλούν ήδη για νέες συνθήκες και η τελευταία συνθήκη ήταν ήδη δύσκολο να την ε, εγκρίνουμε και να αρχίσει να ισχύει, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει βούληση μεταξύ των, πολιτών, των, συμπολιτών μας ε, να αρχίσουμε να μιλούμε για νέες συνθήκες αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι εργαλεία υπάρχουν εντό του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη που ενδεχομένω δεν χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρομαι κυρίω στα πρόστιμα που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα κράτη-μέλη πολύ νωρίτερα και ενδεχομένω να μην είχαμε έτσι οδηγηθεί σε αυτό το επίπεδα ε, χρεών αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρησιμοποιήθηκαν κίνητρα ή αντικίνητρα επίση ε, στο πλαίσιο του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι όταν μιλούμε για κυρώσει. Ε, για γιατί όταν αρχίζουμε να αποσύρουμε ε, πόρους από χώρες που έχουν ήδη μεγάλο χρέος, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακριβώς ακόμη δυσκολότερα και Είδαμε ε, ότι όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση αυτό μπορεί να οδηγήσει αμέσως σε κοινωνική κρίση και δεν πρέπει να μας διαφύγει αυτό. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τι δυνατότητα είχαμε ήδη και μήπως θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον νωρίτερα ως κίνητρο πριν γίνουν τα πράγματα πολύ άσχημα. Όταν έγινε η εξαιρετική ενημέρωση στο ε, Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα με κάποιους εμπειρογνώμονε ε, που μίλησαν για την οικονομική διακυβέρνηση, ε, θα ήθελα να, είχα, ήταν περισσότεροι συνάδελφοι παρόντες γιατί πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη και η δουλειά της γραμματείας και κάποιος από τους εμπειρογνώμονες ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, ε, πιο ανεξάρτητη εποπτεία σε επίπεδο κράτους μέλους. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που σήμερα θα ανακοινώσει τον προπολογισμό του η νέα κυβέρνηση συνασπισμού έχει ε, χωρίσει την αρμοδιότητα για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ε, σε έναν ανεξάρτητο φορέα για τη σταθερότητα ε, του προϋπολογισμού. Επομένως, ε, θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας ε, που θα έχει μία ξεχωριστή θεώρηση της οικονομικής ανάπτυξης και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί και στις υπόλοιπες χώρες μέλη και ήταν κάτι το οποίο ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, ε, για τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και το να εξετάσουμε το γενικό χρέος, νομίζω ότι αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρεται για τους ισολογισμούς και το χρέος, γιατί έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν, βοηθήθηκαν ιδιαίτερα κάποια κράτη-μέλη. Επίσης μιλούμε για την αξιοπιστία των στατιστικών. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία των στατιστικών. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έχουμε πει και σε άλλα φόρα δεν έχει νόημα να ενισχύουμε το σύστημα όταν δεν μπορούμε να βασιστούμε στα αριθμητικά στοιχεία που πρέπει να μας λένε κατά πόσο δουλεύει όχι το σύστημα αυτό. Επίσης, λίγη προσοχή, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα, στη δική μου χώρα, ο εθνικός ε, προϋπολογισμός ε, είναι ε, ο ο ακρογωνιαίος λίθος της κυριαρχίας του κράτους μέλους και αν δεν το λάβουμε αυτό, αυτό υπόψη θα είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα ειδικά για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Σβέν, είχε ζητήσει το λόγο ο Φιλίπ. Πάλι λάθος γράψαμε από τους πρασίνους, ποιος ζήτησε το λόγο. Μερικά σχόλια, ο Φιλίπ Λάμπερτς. Πρώτον, η αμοιβαία εποπτεία. Γίνεται μεγάλος λόγος και δίνεται μεγάλη προσοχή στις δαπάνες, μία διαφωνία. Αλλά θα πρέπει να αντισταθμιστεί αυτό από την εποπτεία και συνεργασία και για τα έσοδα. Βλέπε φορολογία. Είναι δύο τα ζητήματα εδώ. Πρώτον, δεν υπάρχει τρόπος να πετύχει κανείς ισοσκελισμένο ε, προπολογισμό και υγιή με περικοπές και μόνο. Αυτό δεν λειτουργεί ακόμα και εκείνοι που τίνουν περισσότερο να προτιμούν αυτό, ε, ξέρουν ότι δεν πετυχαίνουν. Άρα θα πρέπει να στραφούμε και προς τα έσοδα. Στη συνέχεια, χωρίς συνεργασία δεν υπάρχει τρόπος να επαναφέρουμε ό,τι χάνεται στη φοροδιαφυγή. Γνωρίζουμε, υπολογίζεται ότι είναι 300 δις ευρώ το χρόνο η φοροδιαφυγή και αν θέλουμε ε, να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα στοιχειοδός ή ένα μέρος χρειάζεται συνεργασία με καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από κοινού. Στη συνέχεια επίσης, αν δεν έχουμε φορολογική συνεργασία, τότε η μόνη πηγή την οποία μπορούμε να ε, κυνηγήσουμε είναι ο φόρος εισοδήματος. Ε, και ξέρουμε ήδη ότι έχουμε σφίξει πάρα πολύ το ζωνάρι. Ε, ε, το εισόδημα της εργασίας φορολογείται πάρα πολύ. Θα πρέπει να βρούμε άλλες πηγές λοιπόν που σημαίνει ε, φορολόγηση των συναλλαγών, φορολόγηση των τραπεζών με κάποιο τέλος και ε, με δίκαιη φορολόγηση που ξέρουμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή γεγονός. Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν που σας ζητώ χρειάζεται συνεργασία και κάποιο επίπεδο σύγκλησης του τύπου ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν έχουμε έναν ιαίο συντελεστή, έχουμε όμως ένα περιθώριο όπου μπορούν να κινούνται τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν αυτό το στοιχείο της έκθεσης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Άλλο θέμα. Η κοινοτική μέθοδος απέναντι στη διακυβερνητική. Συμφωνούμε απολύτως. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν θέλουμε να πετύχει η μέθοδος αυτό χρειάζεται συνεργασία και να ενταχθεί μάλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κοινοτική μέθοδο. Αλλιώ θα έχουμε καταστάσει τύπου I want my money back, τα λεφτά μου πίσω που ζητούσε η κυρία Θάτσερ. Και θα αρχίσουν να τσακώνονται διάφορε χώρε μεταξύ του. Τελικά, α, θα πρέπει να συμφωνήσουν και πάλι με του Γερμανού. Και ένα τελευταίο, το στοιχείο τη δημοκρατία, δηλαδή η συμμετοχή κοινοβουλίων. Εκεί θα πρέπει και πάλι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της εμπλοκής των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί σε τελική ανάλυση και για τι δαπάνε και για τα έσοδα και για τη φορολογία η συζήτηση αυτή γίνεται στι εθνικέ βουλέ, αλλά αφού είμαστε ε, στο πνεύμα της κοινοτική μεθόδου πλέον θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σημαντικό ρόλο ε, στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών. Και δεν είναι κάτι λοιπόν που θα επιβληθεί ενιαία σε όλους από πάνω προς τα κάτω το ίδιο. Όχι. Για να βεβαιώσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Τρισέ συνέχεια το αίσθημα του συνανίκην και του κοινού πεπρωμένου κάπου, ότι έχουμε όλη την ίδια μοίρα. Αυτό δεν φαίνεται. Πρέπει να βελτιωθεί κάπως η έκθεση ως προς αυτό το στοιχείο. Κατά τα άλλα έχουμε μια καλή βάση για να εργαστούμε πάνω σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους κοιόδους ε, εισηγητής Κούλ, Κάρινς, Γκότφι uh, Ίνετβελτ, ε, κύριε Κλούτε. Είστε κι εσείς και ο συζητητής, οπότε σε εσάς θα δώσω το λόγο πρώτα, μετά ο Ισβέν και μετά κι εγώ. Κύριε Κλούτε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα. Δύο-τρία μόνο σημαντικότερα. Θέλω να τονίσω κι εγώ ότι έχει νόημα η εποπτεία, αλλά η εποπτεία δεν είναι το παν προφανώς. Υπάρχουν και μηχανισμοί κυρώσεων με μια δική τους εσωτερική λογική, αλλά παρεμβαίνουν στα δικαιώματα κυριαρχίας των κοινοβουλίων των κρατών μελών οι κυρώσεις αυτές. Τουλάχιστον αυτή είναι η θέση της δικής μου πολιτικής ομάδας. Περαιτέρω εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται με υπέρβαση και κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και παραμένει η θέση της ομάδας μου, πάγια. Και κάτι άλλο που δεν αναφέρεται καθόλου. Στο γερμανόφωνο τύπο, επανειλημμένα και εδώ και καιρό, τονίζεται ότι για τα κριτήρια σταθερότητας υπάρχει κάποια μονομέρεια στη συζήτηση, δηλαδή το εμπορικό ισοζύγιο και οι ε, ανισότητες, τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα παίζουν σημαντικό ρόλο και αυτά στη σταθερότητα ε, και δεν το βλέπουμε πάρα πολύ να εμφανίζεται ο κύριος Φλάσπεκ που είναι επικεφαλής του τμήματος ε, παγκοσμιοποίησης και ανάπτυξης της ΟΝΚΤΑ το είπε πρόσφατα. Η ισχύ του ευρώ για τα ασθενέστερα μέλη της ευρωζώνης έχει το εξή αποτέλεσμα. Είναι φτηνές εισαγωγέ και ακριβές οι εξαγωγέ του. Και είναι εις βάρος Αυτό έχει σημασία και οι οικονομίες των ασθενέστερων μελών της Ευρωζώνης έχουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα εξ αυτού και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να αμυνθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Ε, αυτές λοιπόν οι ιστορίες της ανισότητας στο εμπορικό ισοζύγιο θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φέιο για την εισαγωγή του και την παρουσίαση της όσο σημαντικής έκθεσης όσο και επίκαιρη. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ απολύτως με το όραμα που παρουσιάζει ο εισηγητής και συνεχίζει και το ψήφισμα που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με μεγάλη πλειοψηφία για την οικονομική διακυβέρνηση. Πάντως έχει σημασία και στην έκθεση αυτή να τα λέμε και να επεξεργαζόμαστε περισσότερο αυτή την ιδέα οι αρχές που παρουσιάζεται κυρίως για τη λύση με τις 27 χώρες, την κοινοτική μέθοδο, ε, κεντρικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι οι νέα θεσμικά όργανα. Προληπτικά μέτρα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και αυτόματες κυρώσεις. Τα λέτε όλα αυτά. Εχθέ ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριο Τρισέ, μα είπε ενδιαφέροντα πράγματα επ' αυτού και συμφωνούν και με τη δική σας άποψη και θεώρηση. Θα ήθελα και πάλι να το υπογραμμίσω σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Σωστά λέτε ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας και της απασχόλησης. Υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση εκεί, αλλά προσοχή. Να μην είμαστε αμυντικοί στα κοινωνικά θα ήθελα να τονίσετε και μια άλλη πρόπτικη. Όπως και στρατηγική του 2020 θα πρέπει να μιλάμε για κοινωνική συμπερίληψη. Δηλαδή, μια αγορά εργασίας, μια πολιτική που να τονώνει, να αναζωογονεί την αγορά εργασίας και τα κοινωνικά συστήματα, να κινητροδοτούμε δηλαδή την απασχόληση και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ψάχνει δουλειά και να δέχεται τη δουλειά που του προτείνουν. Γιατί η φτώχεια είναι απόρρια της έλλειψης απασχόλησης στην Ευρώπη. Και στις μικρομεσαίες δεν έχουμε θέσει απασχόλησης, γι' αυτό ο κόσμος είναι φτωχός, δεν βρίσκει δουλειά. Και ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε διακυβέρνηση στην οικονομία όχι μόνο για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και στη μικροοικονομικές εξελίξεις. Οι μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Task Force, αυτή την ομάδα κρούσης, με δεσμευτική, γιατί όχι, ισχύει προς τα κράτη-μέλη. Και εδώ συνδέεται με τη στατική για το 2020. Έτσι μπορούμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη στο δρόμο της ανάπτυξης και της απασχόλησης που είναι κρίσιμο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κάρινς, πάνω στην ώρα γυρίσατε. Συγγνώμη, μόλις έχασα αυτά που είπε η, Κάριν. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο είπε χθε ε, και ο κύριος Τρισέ. Είπε ότι υπάρχει ένα παράδοξο. Είπε εν ολίγης ότι χρειαζόμαστε μια ομοσπονδιακή λύση χωρίς ομοστοιχείο ε, ομοσπονδιακό. Κάτι τέτοιο είπε, εν πάση περιπτώσει. Και είναι γεγονός ότι στην οικονομική διακυβέρνηση ισχύει αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι έχουμε μια λύση που να ταιριάζει σε όλους. Η λιτότητα είναι το νέο σλόγγαν ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε οι κυβερνήσει θα μειώσουν ε, τι δαπάνε του για να μπορέσουν να μειώσουν το έλλειμμά του, ε, το οποίο εκ πρώτη όψεω φαίνεται πολύ καλό. Νομίζω όμω ότι. Σε μερικέ χώρες είναι απαραίτητο αυτό και η δική μου χώρα εδώ και 1,5 χρόνο βρίσκεται σε αυτήν τη διαδικασία η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Όλα αυτά πολύ καλά είναι. Ο κύριος Φέγιο ανέφερε επίσης και η κυρία Φόρντ το είπε, πρέπει να σκεφτούμε και την ανάπτυξη. Αν όλοι λοιπόν μειώσουν τις δαπάνες τους, αυτό σημαίνει ότι θα σκοτώσουμε την ε, ζήτηση. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε Μειώνοντα τι δαπάνε, τι θα γίνει με την ανάπτυξη που είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, γιατί αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Είμαι λοιπόν πεπισμένο ε, ότι χρειάζεται ένα κεντρικό συντονιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί να έχουμε σε εθνικό ε, επίπεδο κάτι τέτοιο. Κάθε χώρα θα σκέφτεται την, ε, τα δικά της εσωτερικά ζητήματα χωρίς να σκέφτεται υποχρεωτικά το σύνολο και δεν νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό, υποχρεωτικά ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Ευρωζώνη γιατί ούτως ή άλλως ε, είναι, ε, είμαστε συνδεδεμένοι. Είδαμε τι έγινε με το χρέος της Ελλάδας που επηρέασε και τις χώρες Ευρωζώνης και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Όταν δούμε λοιπόν ε, το πακέτο ε, εργαλείων που έχουμε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τον κύριο Φέη ότι πρέπει να είναι ο κεντρικός συντονιστή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στα μέλη της Ευρωζώνης, γιατί πρέπει, θα ήθελα να τονίσω μία ακόμη φορά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους και μπορεί κάποιος, ε, μπορεί να έχουμε χώρα που ε, εξοδεύει πάρα πολλά και μία χώρα που εξοδεύει πάρα πολύ λίγο. Godfrey Bloom. Πάρα πολύ προσεκτικά άκουσα τους ομιλητές και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που έχουμε συμπεριλάβει και πάλι την ανάπτυξη στο λεξιλόγιό μας. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να το έχουμε ξεχάσει. Ο μόνος τρόπος να βγούμε από το λάκο που έχουμε σκάψει είναι η ανάπτυξη. Και θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση για την ανάπτυξη. Μόνο δύο είδη ανθρώπων υπάρχουν. Υπάρχουν εκείνοι που δημιουργούν πλούτο και εκείνοι που ε, τον ξοδεύουν. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλούς ε, ε, στο δημόσιο τομέα. Υπερβολικά πολλούς. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω για τις υπόλοιπε χώρες, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε φιλανθρωπίες, έχουμε περιφερειακές αρχές, έχουμε δημόσια χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες, έχουμε πράσινη Θέσει ε, θέσεις απασχόλησης ε, που καλύπτουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί δημιουργούν πλούτο ε, και δεν είναι υποχρεωτικά κάτι που καταλήγει σε αύξηση, των, σε, ανάπτυξη και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά σε χώρες με, μικρότερες, με μικρότερο δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, κάνει τίποτε γι' αυτό. Εμείς είμαστε, πρόβλημα, είμαστε τμήμα του προβλήματος και όχι της λύσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να ακούσω τον εισηγητή. Έφτασα καθυστερημένο. Καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα κείμενο το οποίο έχει κυκλοφορήσει αλλά δεν έλαβαν όλοι Εγώ σαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πραγματικά δεν είμαστε φαίνεται όλοι σε ίδιο επίπεδο ισότητος. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, η οποία έρχεται σε ένα σημείο, σε μια διαδικασία αποφάσεων, η οποία έχει ξεκινήσει και πιστεύω, κυρία Βόρτμαν Κόλλ είχε δίκιο όταν είπε προηγουμένως ότι τα ψηφίσματα που είχαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα πλαίσιο σε αυτή την έκθεση. Εάν θέλουμε να είμαστε συνενετικοί για το πέρας της κρίσης, για το πόσο που θα πρέπει να βγάλουμε για την κρίση. Το σημείο εκείνη σύγκληση είναι η συμβολή της Κομισιόν στην ομάδα εργασίας που, που προεδρεύεται από τον Φόνον Πόη. Αυτό είναι το σημείο κίνησης και εφόσον έχουμε την έκθεση αυτή που ξεκινάει θέλω να κάνω μεθοδολογικό στοιχείο, να υποβάλω μάλλον. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, ωστόσο πάσχουν μιας μίξης των διαφόρων ειδών, δηλαδή τα μέτρα αφενός και τα πολιτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και αυτά τα δύο επειδή αναμειγνύονται κάνουν τα πράγματα πολύ πιο περίπλοκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σήμα θα δώσει ένα σήμα με βάση την απολογισμό της λειτουργίας του ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και από αυτή τη σκοπιά μερικοί ανακαλύπτουν ορισμένα στοιχεία με βάση αυτή την κρίση που περνάμε. Αυτά είχαν λεφθεί και παλαιότερα και λεγόταν ότι υπάρχει μία διαφορά της ανταγωνιστικότητας και ότι μία δεν υπήρχε σύγκληση αλλά απόκληση. Είναι ένα φαινόμενο για το οποίο ελέγχθη ότι το, το, ε, το πρωτόκολλο για τη σύγκληση και την ανάπτυξη δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο το οποίο χρειαζόταν. Πρέπει να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή η ζώνη ευρώ πρέπει να δούμε το σύμφωνο αυτό ξανά από την αρχή. Χρειάζεται ένα σύμφωνο το οποίο θα είναι ισχυρό, αλλά δεν θα είναι το βασικό στοιχείο της συζήτησης. Το πρώτο στοιχείο θα είναι πώς θα καταπολεμήσουμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν, πώς θα, υπά... θα συγκρίνει αυτή η διαφορά μεταξύ εξαγωγέων και εισαγωγέων, πώς θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο, ούτως ώστε με βάση το κοινό συμφέρον της κοινότητας, όπως το είπε και ο Λιμό θα, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό το στοιχείο το οποίο θα συμβάλλει περισσότερο, περισσότερο στην σύγκληση. Τώρα θέλω σε ένα σημείο το οποίο είναι θεσμικό. Ξέρετε όσον αφορά την κρίση είχα κάνει μια πρόταση η οποία συζήτηκε τότε στο, συντακτικό όσον αφορά το Σύνταγμα και θα έπρεπε είχα πει να βρούμε τον τρόπο για να εξετάσουμε ποια είναι η ιδέα ότι δεν υπάρχει μία, μία διαχωριστική γραμμή, ένα τείχος μεταξύ των 27 και των 16, 16-27 και ότι υποχρεώνει και τις ε, οι 16 αποκλειστικά έχουν μια ευθύνη περισσότερη γιατί έχουν το ευρώ. Τι αυτή είναι η διαφορά. Αλλά βλέπετε εδώ και 12-13 χρόνια τα πράγματα λειτουργούν. Δεδομένου, ότι αυτοί που συνέταξαν το Μάστριχ είχαν ένα πρόβλημα το οποίο δεν το επέλυσαν. Και αν δεν το επιλύσουμε θα συνεχιστεί και η κρίση. Ότι νόμιμα αυτή τη στιγμή η πολιτική, η πολιτική των προϋπολογισμών των κρατών μελών και η νομισματική πολιτική είναι της Ευρώπης. Εάν δεν ξεπεράσουμε αυτό το βασικό θέμα κλειδί, εάν η Κομισιόν ασχολείται, ασχολείται για τα πάντα και απλώς τα κράτη κάνουν ό,τι τους κατέβει, δεν θα προχωρήσουμε ούτε σπιθαμή. Πιστεύω λοιπόν αυτό το πράγμα θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα τομέα όπου υπάρχουν αρμοδιότητες που είναι διχασμένες. Όλοι φωνάζουν, τσιρίζουν και λένε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμό. Αλλά ο συντονισμό δεν μπορεί να την κάνει η Κομισιόν, που είναι παντοδύναμη τάχα μου. Θα πρέπει επί του ιδίου μοντέλου, όπω η κυρία πολιτική εξωτερική πολιτική όπως έχουμε θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο ο οποίος θα είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν ε, ε, και ο οποίος θα έχει την νομιμότητα και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να προχωρήσει αυτό το θέμα που σας ανάφερα. Δύο λεπτά ακόμη Πρόεδρε. Θεσμική πτυχή όσον αφορά τη συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων. Το κοινο... Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κύκλος για αυτό το θέμα. Αλλά ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή τη στιγμή ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα παραδεχθούν τη μεταφορά του προπολογισμού από την αρμοδιότητά τους. Δεν θα το δεχθούν αυτό το πράγμα. Θα είναι αντικυκλικό αν θέλετε. Πώς αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια απόφαση η οποία θα είναι εκτός, εκκεντρική εκτός του κέντρου και πώς ακριβώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κοινοβούλια και πώς ακριβώς αυτά τα, τα, ε, τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια των χωρών μελών θα πρέπει να συνάδουν με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θα είναι πιο ευνοϊκός. Στη συνθήκη σήμερα αυτή τη στιγμή όταν ένα κράτος ε, ε, υφίσταται κυρώσεις δεν συμμετέχει στις συναποφάσεις. Αυτή η διάταξη έχει ληφθεί και είναι λογικό. Αλλά η κατάργηση του δικαιώματος του, ψηφί, του ψηφίζει είναι παράλογο διότι κάποιος όταν μπαίνει στην ΕΕ ψηφίζει βασικά και δεν καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει όταν γίνουμε μέλος της, Ευρω... Ευρωζώνης τότε μας καταργεί το δικαίωμα του της ψήφου Νομίζω πως το θέμα της δημοκρατίας μου φαίνεται ότι είναι το μείζον θέμα. Εάν καταργήσουμε την ψήφο λοιπόν πιστεύω πως είναι συμβολικά και αντιπαραγωγική αλλά και πολύ βαριά και αντιδημοκρατική αν θέλετε. Εάν θέλουμε να υπάρχει σύγκληση ευρωπαϊκή λοιπόν θα πούμε «Α, θέλουμε σύγκληση αλλά σκάσε, συγγνώμη για την έκφραση, μη μιλάς, βούλωσέ το, εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε και δεν έχεις και δικαίωμα ψήφου». Σας καλώ λοιπόν να το διευρύνετε. Θα υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες είναι έξυπνες. Για παράδειγμα, μια χώρα η οποία μπορεί αυξάνεται το ΦΠΑ, αυξάνεται το φόρος επί των καυσίμων, αλλά κυρώσεις, κυρώσεις οι οποίες κάνουν τον άρρωστο να αιμορραγεί. Δεν είναι κυρώσεις αυτές, είναι αντιπαραγωγικές. Αυτό προτείνουμε εμεί στην πρόταση. Συγγνώμη, μακρηγόρησε. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ, Περβάς. Μάλλον θα έχουμε χρόνο στο τέλος τη ψηφοφορία, Η Σόφι Νετβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να μην πάρω πολύ χρόνο από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ την ίδια παρατήρηση με την Περβάς. Θα ήταν πιο εύκολο να συζητήσουμε αν είχαμε λαβεί όλοι προηγουμένως το έγγραφο. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά ζητήματα. Επί της προσοχή να μην δημιουργήσουμε στρεβλή αντίφαση μεταξύ της ανάγκης δημοσιονομικής πειθαρχία και ανάπτυξης. Γιατί οι δημόσιες δαπάνες δεν ταυτίζονται απαραίτητο με δημόσιες επενδύσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή όταν έχουμε περισσότερες δημόσιες δαπάνες ότι θα είναι επενδυτικές αυτές οι δαπάνες με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για την ανάπτυξη επίσης δεν έχω ακούσει ακόμα, αλλά μπορεί να είμαι και αφηρημένη, ε, πώς θα αυξηθεί η ε, παραγωγικότητα, με επενδύσεις στη γνώση, πιο ευέλικτη αγορά εργασίας και να μην προστατεύει τα προνόμια των εργαζομένων αφήνοντας εκτός αγοράς εργασίας άλλους που θέλουν να εργαστούν. Συγγνώμη. Δεν άκουσα πάρα πολλά ε, επίσης για το πώς θα ολοκληρωθεί περισσότερο η εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες. Συνέχεια για κρατικές δαπάνες μιλάμε. Γιατί αποφεύγουμε να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις. Ε, δεν θα πρέπει να τα συζητάμε και αυτά καμιά φορά. Και μετά, για τη μέθοδο. Με μεγάλη προσοχή άκουσα αυτά που είπε η κυρία Φόρτ. Και παρόλο που πρέπει να σας πω ότι ε, τα βλέπω με συμπάθεια και κατανόηση και αναγνωρίζω αυτά που λέτε, οι περισσότεροι ψηφοφόροι μας αρνούνται και νέα εκχώρηση δικαιωμάτων και κυριαρχίας προς τις Βρυξέλλες. Έχουν μπουχτίσει πλέον. Και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα ήταν βασικά συμφωνία κυρίων ε, να μην παρεμβαίνουμε ο στα χωράφια του άλλου. Και δεν δούλεψε, ούτε πρόκειται ποτέ να δουλέψει. Όσο και αν επαναλαμβάνουμε ότι οι κυρώσει θα πρέπει να επιβάλλονται, γνωρίζουμε όλοι ότι τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, λέγω, που θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσει το ένα στο άλλο, δεν θα το κάνουν. Επίση, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν όλα ίση μεταχείριση. Γιατί όταν βγαίνει στη Γερμανική Βουλή η κυρία Μέρκελ και λέει εάν δεν τηρήσει τι υποχρεώσει τη η Ελλάδα, τότε ίσω θα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη. Δεν φαντάζομαι να πει ακριβώ το ίδιο για τη Γαλλία η κυρία Μέρκελ, αν δεν τηρήσει τι υποχρεώσει τη η Γαλλία στο καλό από την Ευρωζώνη. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό στα χέρια των κρατών μελών να επιβάλλουν κυρώσει το ένα στο άλλο διότι ποτέ δεν πρόκειται να το κάνουν, απλούστατα. Κοιτάξτε, άλλο τομέα πολιτική, το άρθρο 7, που αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, τιμωρήσει ένα κράτος μέλος... Ε, και σε πολλέ περιπτώσει θα μπορούσε να το είχε κάνει, δεν το έχει κάνει, να αναστείλει τη συμμετοχή ενό κράτου, α πούμε, στα όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπόλογοι και στους πολίτες και εκείνοι θα πρέπει να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και ένα τελευταίο. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίε. Πρόεδρε, γίνεται πολύ φασαρία στην αίθουσα. Συνάδελφοι, συζητήσετε η συζήτηση και ίσως θα μας έκανε καλό, λέει η Πρόεδρος, σε όλους να ακούμε. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Νετβέλτ, τώρα. Έλεγα λοιπόν, για το ε, εκ των προτέρων έλεγχο των εθνικών, των κρατικών προπολογισμών και πώς μπαίνει στα χωράφια της κυριαρχίας. Όλα αυτά ισχύουν και είναι σωστά. Αλλά δεν άκουσα ακόμα καμία συζήτηση για την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων. Ποια είναι η ευθύνη τους, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα για το ε, σταθερότητα της Ευρωζώνης τίποτα. Μηδενική ευθύνη. Κοιτούν μόνο τα εθνικά του συμφέροντα. Και βέβαια, ίσω να μην μπορεί κανεί να περιμένει περισσότερα από εθνικά κοινοβούλια. Αλλά να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Όταν θε εξουσίε, οι εξουσίε συνοδεύονται από ευθύνε και θα πρέπει να τι αναλαμβάνουν. Αν δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του, τότε α μην έχουν και τι εξουσίε τα κοινοβούλια. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ισχυρή οικονομία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι περισσότερο από 27 φορές ε, εθνικά συμφέροντα. Και δεν είμαστε σε κανένα νησί, όσο και αν το νομίζουμε, αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Και συμφέρει τους ανταγωνιστές μας να είμαστε διχασμένοι και αδύνατοι. Θέλουμε να είμαστε ενωμένοι ως Ευρώπη. Θέλουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί χρειάζεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Επειδή έχει προχωρήσει η ώρα, θα ήθελα να τονίσω μόνο ουσιαστικά ένα σημείο. Στη συζήτηση αυτή νομίζω θα πρέπει να έχουμε λίγο την αίσθηση του κατεπήγοντος και να προσέξουμε να μην χρησιμοποιήσουμε την ίδια διατύπωση με εκείνη που κάναμε για την Ευρωζώνη. Τώρα είμαστε σε άλλο στάδιο της κρίσης, σε άλλη φάση της κρίσης και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στα μέτρα που υποστηρίζουμε και στο βάθος των μέτρων που υποστηρίζουμε. Θα ήθελα, και πάλι γίνεται μεγάλη φασαρία πρόεδρε στην αίθουσα, θα ήθελα να τονίσω θα ήθελα να τονίσω λέγω την ανάγκη να μην αποφύγουμε τη συζήτηση. Και υπό την έννοια αυτή συμφωνώ και με αυτά που είπε η Σόφη. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη συζήτηση ή τις συζητήσεις στο πληθυντικό για ε, τις μεγάλες ανισότητες ε, της οικονομίας και τις ευρωστίες της οικονομίας σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Θυμάμαι πολύ καλά στην έκθεση για την Ευρωζώνη ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να αφήσουμε στην άκρη όλες τις πρακτικές ε, ε, υποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και ε, τις ανισορροπίες. Και τώρα βρεθήκαμε ε, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χάος. Δεν μπορεί απλώς να λέει η πλειοψηφία, η πλειοψηφία ότι δεν μπορούμε να δράσουμε εδώ και θέλουμε επιπλέον κριτήρια στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αλλά χωρίς πρακτικά μέτρα που να εφαρμόζονται για να φτάσουμε στη σύγκληση. Χωρίς σύγκληση η Ευρωζώνη ε, τουλάχιστον θα αποτύχει. Και ως κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό πέρα από την οικονομική φιλοσοφία του καθενός. Αυτή τη φορά πιστεύω θα πρέπει να είναι σκληρά τα επιχειρήματα ε, κατά της αδράνειας και υπέρ των πρακτικών μέτρων. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό για μερικές πολιτικές ομάδες και ορισμένες από τις προτάσεις να είναι πολύ ιδεολογικά φορτισμένες, πολύ δύσκολο να τις δεχτούμε, αλλά δεν μπορούμε τώρα ξανά να αποφύγουμε, να προτείνουμε πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση ε, για την ανταγωνιστικότητα, για τις ανισορροπίες. Ξέρω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για τον συγητή να καλύψει τα κενά, να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων αλλά και περιφερειών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. I... Ευχαριστώ. Λυπάμαι. Ε, ε συγγνώμη, που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω μερικά σημεία και θα πρέπει να σταματήσουν τον κατάλογο. Το κείμενο το κείμενο που παρουσιάστηκε και το οποίο ασπάστηκαν εν μέρη και μίλησαν οι ο ομιλητικής, νομίζω θα μιλήσουν και άλλοι και θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ αυτό το πράγμα και θα πρέπει να είμαστε προκλητικοί. Και όπως είπε και στις εχθές, θα πρέπει να πάμε όσο γίνεται στα πλαίσια της παρούσης συνθήκης, όσο μακριά μπορούμε. Αυτό θα δώσει το ΜΑΚ ε, με το 126 σημείο 6 και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πάει όσο μακριά γίνεται σε αυτό το θέμα, στα όρια της συνθήκης δηλαδή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός ο οποίος θα οδηγεί βεβαίως σε μια πειθαρχία επί του προλογισμού αλλά θα πρέπει να έχουμε καλύτερο έλεγχο των στοιχείων της Eurostat και θα πρέπει μεταξύ αυτών να γίνεται ένα συντονισμό μεταξύ κρατών μελών για να μην υπάρχουν αυτά τα οποία είχαν προηγουμένως και μην υπάρχουν φθόρες διαρροές αν θέλετε και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλον. Όπως είπε και ο Τρισιάκομι χθε, θα πρέπει να δούμε ε, έναν αυτοματισμό ή, ή μη αυτοματισμό. Δηλαδή τα πράγματα ή θα γίνονται με αυτό το μία αυτόματο τρόπο ή δεν θα γίνονται καθόλου. Και ε, βεβαίω υπάρχει μια αντίθεση εκ μέρου των αγορών. Αυτό είναι για τον οποίο υπάρχει μια οδηγία όσον αφορά ε, την το κεφάλαιο και τι ακριβώς σχέση έχει αυτό με το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο δανεισμό. Αυτό είναι ο αυτόματος είπε, αλλά υπάρχει για τον αυτόματο τρόπο έλεγχο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι πολιτικό, το οποίο περνάει και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Δεν είναι η Κομισιόν η κακή και το Συμβούλιο το καλό το οποίο τα αφήνει εκτός ημερήσιας διάταξη μερικέ φορές. Νομίζω πως υπάρχουν πτυχές οι οποίες είναι δύσκολες και είναι κύριες οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται πολύ περισσότερο από την αγορά. Νομίζω θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι χωρίς να υπάρξει αλλαγή της συνθήκης βεβαίως, αλλά να φτάσουμε στο όριό μας και να δώσουμε ένα νόημα το οποίο θα έχει μία επίπτωση σε μία μεγάλη χώρα βεβαίως. Ίσως η κυρία Μέρκελ σκέφτηκε, και, σκέφτηκε κάτι και νομίζω πως αυτό το πράγμα υποστηρίζει. Αυτά ήθελα να πω και δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή εάν θέλει κάτι να προσθέσει. Λίγο λυπάμαι που καθυστερήσαμε την ψηφοφορία αλλά είχαμε αυτό το χρόνο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα υποβάλω καταρχήν τις ευχαριστίες μου. Όλοι οι συγητές, οι, οι σκιώδεις, θα, θα, θα πρέπει να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς και όλους αυτούς οι οποίοι παρενέβησαν σήμερα στη συζήτησή μας. Έλαβα πολλές σημειώσεις, σελίδες ολόκληρες σημειώσεων γνωρίζετε είμαστε ήδη καθυστερημένοι. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή όλες τις παρεμβάσεις. Ωστόσο θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Η μέθοδος στην οποία αναφερθήκατε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η προθεσμία και το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σφιχτό. Δεν έχουμε χρόνο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξ αποφάσισα να μοιράσω το κείμενο κείμενο επί του οποίου εργάστηκα και να το δώσω σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές για να μπορέσουν να, έχουν, να έχουμε μάλλον τις απόψεις των διαφορών πολιτικών ομάδων επί των θεμάτων τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα. Αυτό το έκανα για λόγους αποτελεσματικότητας βεβαίως. Το, το μοίρασα το διένυμα αυτό το κείμενο σε όλους κατά τη διάρκεια της εξάρτησης των όλων φάσεων της εξέλιξης της εκθέσεως για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε για ένα κείμενο το οποίο, το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι και υπάρχουν βεβαίως συμμορισμένοι εντό της θεσούς αυτής οι οποίοι δεν αρέσκονται σε αυτό το κείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Το κείμενο λοιπόν θα μεταφερθεί, θα σταλεί το τέλος αυτής της εβδομάδας και στο Στρασβούργο θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Δύο ακόμη σημεία. Αυτό το κείμενο είναι ένα κείμενο συνέχειας ε, άλλων κειμένων τα οποία παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε τι είχαμε παρουσιάσει, τι είχαμε υιοθετεί στο, στο Στρασβούργο όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης και εδώ δεν έχω εγώ σκοπό να κάνω ένα κείμενο το οποίο θα έχει ιδεολογική βάση επί διαφόρων θεμάτων απλούστατα επιθυμώ να εγγραφώ σε ένα πνεύμα στο πνεύμα του άρθρου 3 της συνθήκης το οποίο ορίζει σαν στόχο της Ένωσης την ανάπτυξη, την ισορροπημένη ανάπτυξη της ΕΕ, μια ισορροπία των τιμών, μια ανταγωνιστικότητα που θα είναι υψηλού επίπεδου και το οποίο θα οδηγήσει στην πλήρη απασχόληση και στην κοινωνική ανάπτυξη. Αυτή ήταν η στόχη επί των οποίων εγώ επιθυμώ να εργαστώ και ακόμη μια φορά επαναλαμβάνω και επιβεβαιώνω πως θα πρέπει να κάνουμε μια ευκαιρία από αυτή, να βγάλουμε μια ευκαιρία, να μας δοθεί μια ευκαιρία από αυτή την κρίση και επιμένω σαν εισηγητή και λέγω πως θα πρέπει να φτάσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη συνενέση που μπορούμε σε αυτά τα θέματα με όλες τις πολιτικές ομάδες ούτω ώστε να καταστεί δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακουστεί προς τα έξω με ένα συνενετικό τρόπο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβολές σας όλους. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μία παρουσίαση του, σχεδίου έκθεσης της 5 Ιουλίου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 7 Σεπτεμβρίου. Εξέταση τροπολογιών 27 Σεπτεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 4 Οκτωβρίου και ελπίζουμε για την Ολομέλεια πάλι του Οκτωβρίου. Συγγνώμη που σας τα λέω έτσι μαζεμένα. Αλλά θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει το σχέδιο έκθεσης εγκαίρως μαζί με την νομοθεσία και γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να βιαστούμε λιγάκι. Υπάρχει μία συζήτηση ανοιχτή των συντονιστών με την ομάδα εργασίας ε, του Φαν Ρόνπαϊ ε, στις 30 ε, Ιουνίου. Θα σας πούμε λεπτομέρειες αργότερα. Όσοι λοιπόν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει στην Task Force, σημειώστε την ημερομηνία αυτή στην ατζέντα σας. Λοιπόν, δεν χρονοτριβούμε άλλο. Παρακαλούμε βάλτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας ε, στη σχισμή για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε υπεράριθμους. Αν έχουμε λίγους, τι να πω, τόσο το χειρότερο. Έναρξη δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Δουλεύουν οι κάρτες όλων. Κύριε Κάρας. Έχετε την παλιά σας κάρτα. Μάλιστα. Ε, okay, but if we if, if... Αν ε, είναι πολύ τσιματσίμα η ψηφοφορία, θα δούμε. Ε, πώς θα λάβουμε υπόψη ε, κάποιες, ε, κάποιες επιπλέον ψήφους. Λοιπόν, περνάμε στην έκθεση της κυρίας Φερέιρα για την διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στο τραπεζικό τομέα. Συμβιβαστική τροπολογία Α, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1, υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική B υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική E. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Μερικές σελίδες μετά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική G στη σελίδα 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Σελίδα 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 1 υπέρ Α, όλες οι αιτιολογικές αναφορές θα τις ψηφίσουμε μαζί. Μέχρι τη 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Αιτιολογική σκέψη 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 11α νέο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όλες μαζί μπορούμε να τις ψηφίσουμε μέχρι το τέλος ε, των ε, αιτιολογικών σκέψεων. Μέχρι τη συμβιβαστική Α, υπέρ. Όχι. Λοιπόν, τότε μία-μία. 13 η αιτιολογική αναφορά 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια για την αιτιολογική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας ε, για την EA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη FC νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. FC New και πάλι υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. γρομοδότηση της, νομι... Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, αιτιολογική σκέψη FC νέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Και ο κύριος Κάρας έβαλε την κάρτα του. Η δική μου δεν δουλεύει όμως. Α, ε, όχι, δουλεύει. Δεν μπορώ να ψηφίσω όμως. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Χωρίς τη δική μου βοήθεια. G, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Μπορούμε να ψηφίσουμε την αιτιολογική σκέψη G. Έναρξη ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικής. Η δική μου κάρτα εξακολουθεί να μην δουλεύει. Ο εδώ ψηφίζει για μένα. Ενδιαφέρον. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πού είχαμε φτάσει? Λοιπόν, αιτιολογική σκέψη H, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. A, νέα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη I με προφορική τροπολογία τη ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 καταπίπτει. Οπότε σκέψη IA νέα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. IB νέα υπέρ κατά. Αλλά θα πρέπει να το ελέγξουμε την αιτιολογική σκέψη IB νέο κείμενο. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η πλειοψηφία σήμερα είναι 23 ψήφοι. Συμβιβαστική εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχηγό κείμενο K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική σκέψη L. Τροπολογία... Α, μόνο το αρχικό κείμενο πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. KB με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NB νέο, ναι, όχι καταπίπτει αυτό. Συμβιβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται PA νέα με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τρεις ακόμη μένουν να ψηφίσουν. πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και συνεχίζουμε. 8. Και άλλη ψηφοφορία Τη έκθεσης κυρίου Ελχαντράουη. καθεστώ αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιριών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι. Όλοι. Η τροπολογία περιφών 14. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Είστε όλοι μαζί μου. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο πολύ την ώρα που ψηφίζουμε. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτεται μεταξύ των ψηφισάντων 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 16 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί θέλετε έλεγχο αν θέλετε βεβαίως ωραία ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 16 παρακαλώ αρχίζει ψηφοφορία στην τροπολογία 16 βρισκόμαστε. 16! Ένα, 6! Δική σου τροπολογία είναι, Κάρλα, που ρωτάς κιόλας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική α, ψήφι π, κατά. Ορίστε. Μια στιγμή, γιατί έχουμε κατατμήματα εδώ. Ωραία. Εδώ λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα το υπόλοιπο κείμενο. Το υπόλοιπο κείμενο ε, ψήφι υπέρ είναι το πρώτο τμήμα, κατά αποχές κλπ. εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Και προχωρούμε. Στην 20. Ψήφι υπέρ της 20 κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική Β, και πάλι κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τσεκ. Το ΕΛΚ κάτι ψήφισε ή άλλη τίποτα. Μπορούμε να ψηφίσουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασα. Τώρα εγκρίνεται. Τώρα εγκρίνεται, βάση περιπτώσει. 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Την 24 λοιπόν ελέγχουμε αρχής ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Right, vote's closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ορίστε. 30-17. 25. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Ψήφι π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική ε, C όλοι μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και ερχόμαστε στην 38, αν δεν απατώμε έτσι. Δυστυχώς δεν γράφει εδώ η λίστα που πρέπει να πάω. Στην D η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στην 38. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 της ε, ε, απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 43 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές α, συγγνώμη, τώρα είμαστε στη 45 θα επανέλθουμε 44, την ξέχασα λοιπόν, ε, είμαστε στη μέση της 45 τώρα, να συνεχίσουμε υπέρ της 45 κατά 45 θα έρθουμε και στη 44 κατά αποχές απορρίπτεται τώρα η 44 είναι συμβατή με τη 43 Υπέρ τη 44 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μα πέρασε η 43. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Έτσι δεν είναι. Θέλεις έλεγχο για τη 44. Ωραία, στην ελέγξουμε τη 44. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την 44 παρακαλώ. Ψήφισαμε όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 17 υπέρ, 26 κατά. Δίκιο είχα. Λοιπόν, η 45 έχει απορριφθεί και τώρα θα ψηφίσουμε τη 46 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα το αρχικό κείμενο της παραγράφου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 και 48 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 6 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 συμβατή ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σηκώσατε χέρια. 51 την ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Αγκρίθηκε. Λοιπόν, ήταν ε, προφανής η έγκριση. Ε, πάμε στην 53. Ψήφι Π. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 54 Π. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 και 56 μαζί πε, Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. 55 και 56 μαζί ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 28-19. Διαγράφεται κτλ. Προχωρούμε. Συμβαστική ε ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δυνάμει σελίδα. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα η Τρία τροπολογία. ψήφιπε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα 64, κατά τμήματα, τμήμα πρώτο, το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα για το 50% Αν υπερψηφίσετε σημαίνει ότι είστε υπέρ του 50%. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται λοιπόν το υπόλοιπο κείμενο εκτός του τμήματος 2 που βλέπετε γραμμένο εδώ. Και τώρα θα πρέπει να πάμε στην 65. Είχα προχωρήσει εγώ, αλλά όχι. Είστε σίγουροι ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 65, δεν καταπίπτει. Καλά. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα 67. Προχωρήστε μέχρι την 67. Είναι και η δική μου και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγωση 7 της απασχόλησης. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 επε κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται επίση. Η παράγραφος 11 της απασχόλησης ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 16 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 της Επιτροπής Απασχόλησης Είπε κατά αποχές απορρίπτεται. 69 τροπολογία Είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 είπε Θέλετε έλεγχο για την 69. Καλώς, ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά, την 69. Κοιτάξτε κάτι περίεργου αντίχειρε που σηκώνονται εδώ. Λοιπόν, εγκρίθηκε. Η εννέα της αποσχόλησης υπέρ. Κατά. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε λίγο σας παρακαλώ. Η εννέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 2 της απασχόλησης ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 είπε. Κατά. Αποχές. Είναι περίεργο σύγχυση προκαλεί. Ας το ελέγξουμε όμως. 81 τροπολογία παρακαλώ. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ε, εγκρίθηκε. 17 καταπίπτει λοιπόν, συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 15, παράγραφος 15 της απασχόλησης. Τι λέει εδώ. Ναι, υπέρ της 15 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, αιτιολογικές αναφορές. Α, συγγνώμη, έχουμε και στην παράγραφο 28 το αρχικό κείμενο. Δεν ήταν η ίδια παράγραφο. έκανα λάθο. Είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα στι αιτιολογικέ αναφορέ. Ε, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5α νέα υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η αιτιολογική αναφορά 6α νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6c υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα αιτιολογικές Αλφα κάτα ε, από σχέσει εγκρίνεται. υπέρ τη α κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ τη προφορικη κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 4, ε, συγγνώμη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά Ζων Πολ ψηφίζεις ξανά την 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται β της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία νέα. Όχι, όχι μια στιγμή. Αιτιολογική σκέψη C της απασχόλησης. Αιτιολογική σκέψη C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η νέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η νέα αιτιολογική αναφορά υπέρ κατά σκέψη, συγγνώμη, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, 10 και 11 τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία παρελθόν 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο τώρα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Yeah. Hang on, we're in the middle of a vote. Have you got a problem? Είμαστε στη μέση ψηφοφορία. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Τι έγινε? Πέρασε. Εγκρίθηκε. 40. Ποιο θέλει το λόγο? Ήθελα να κάνω επεξήγηση ψήφου. 30 δεύτερα στον εισηγητή. Καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή παρά τις πρόοδους, ορισμένες πρόοδους που έχουν γίνει, γιατί η αλλαγή ψηφοφορία στην παράγραφο 18 ε, φέρνει την έκθεση αντίφαση ε, με το όσα ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν είναι πολύ υπέρ του ειδικού μας βάρου στον τριμερή διάλογο, γι' αυτό καταψηφίσαμε το λόγο την έκθεση αυτή. Η πρόεδρο. Ελπίζω να μην επηρεάσει πάρα πολύ αυτό τη στάση μας στο τριμερή διάλογο. Προχωρούμε στο σημείο 8. 8 ήμασταν τώρα. Σημείο 9. Σήμερα, ναι, λοιπόν, είστε όλοι παρόντες εδώ, μια χαρά, πάμε. Η πρώτη ψηφοφορία, unblock, η συμβαστική λύση, η οποία προπολογία που η ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, Unblock στο σύνολο, στο συμβαστική λύση, στο κείμενο στο οποίο υπάρχει. Ψήφισαν οι πάντες. Όχι ακόμη. Πέρας. Υιοθετείτε. Τώρα πάμε. Όχι. Θα ψηφίσουμε το σύνολο όχι. Ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία για την νομοθετική πλευρά του κειμένου. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Υιοθετείτε. Μία ψήφος κατά μόνο. Συγχαρητήρια. Κύριε Μπινεύ. Λαμπρά. Τελειώσαμε πολύ γρήγορα με το κείμενό σας. Πάμε τώρα. Σημείο 10. Στο σημείο 10. Ε, προφορική ερώτηση όσον αφορά, που θα έρθει στο επόμενο Στρασβούργο όσον αφορά το μηχανισμό ε, χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης και στις μελλοντικέ δράσεις. Θα πάει με τις παραγράφους. Παράγραφο 1 είναι υπέρ, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική λύση 2, ως κατά αποχές υιοθετείται. Ερχόμεθα τώρα το σημείο, σημείο 3 ο συνυπέρ κατά αποχές υιοθετείται 3α υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 4α υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως υιοθετείτε, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 4α. Ηλεκτρονικός έλεγχος πάρτε τις κάρτες σας. Ψήφισαν οι πάντες. Σιλβί. Ναι. Ναμπρά. Πέρας. Υιοθετείτε. Με μία ψήφο μόνο. 23-22. 4β υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 5α υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 5β υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. ηλεκτρονικά τώρα όπως τοποποιήθηκε το κείμενο με τις κάρτες σας παρακαλώ Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Συμφωνούμε απαξάπαντες. Πλήρης ομοφωνία. Λαμπρά. Ερχόμεθα τώρα. Πάμε, δεν πάμε, πάμε. Λέει πρόεδρος. Σικλούνα, ανάπτυξη του νοικομικού δημιουργία θέσεων εργαστικό στο πλαίσιο μια βιώσιμη οικονομία. Ένα. Δύο. Υπέρ κατά αποχέ υιοθετείτε. Συμβαστική Α. Υπέρ κατά αποχέ υιοθετείτε. Νομίζω ότι υιοθετείτε. Ναι. Ναι, μερικοί ψήφισαν αρχικά. Β. Συμβαστική υπέρ κατά αποχέ υιοθετείτε. τρία υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 5 υπέρ α μετική ψηφοφορία πρώτο σημείο ως πρώτο υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται επίσης τοπολογία 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 7 υπέρ κατά μια στιγμή χωρίς μικρόφωνο κάποιος παρεμβαίνει η πρόεδρος η τροπολογία αντικαθιστά την τιματική ψηφοφορία έτσι το αντιλαμβάνεστε μπορεί ο εισηγητής να επιβεβαιώσει αυτό που λέω έτσι δεν έχουν τα πράγματα να μπρά Παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 9 ναι, τροπολογία υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ στο κείμενο έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή λαμπρά Πέρασε ψηφοφορίες, ομόφωνα συγχαρητήρια στον εισηγητή τελική ψηφοφορία σήμερα το πρωί ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία που είναι του Hans Peter Mitt Martin κατευθύνει γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών ε, συμβαστική α κατά υπερ Παρακαλώ να ελέγξουμε την α, συμβαστική λύση α, ηλεκτρονικά. Ψήφισαν οι πάντες, πέρας. Υιοθετείτε. εξτροπολογία, δύο μέρη, πρώτο μέρη, ε, 46 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Απερίφθη, συγγνώμη, 46. Στο δεύτερο σημείο του 46 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε λέει πρόεδρος διακόπτοντας. Σημείο 46 β, δεύτερο σημείο, το δεύτερο μέρος, ψήφισαν οι πάντε, πέρας, απερίφθη. 47 ψήφισαν οι πάντε ε, ψη, υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να το ελέγξουμε το 47 47 ψήφισαν οι πάντες πέρας απερίφθη το 47 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Οκτώ. υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά το, την συμβαστική πρόταση β Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας και υιοθετείτε. Ναι, υιοθετείτε. 50 τοπολογία. 50. Όλε Λούτφιξον υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. Συμβαστική πρόταση γάμα, Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 53 το τροπολογία υπέρ κατά αποχές νομίζω πως θα περιευθεί αλλά θα το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά 53 ψήφισαν οι πάντες πέρας απεριφθεί όντως 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 55 υπέρ κατά να το ελέγξουμε γιατί δεν ξέρουμε ποιοι ψήφισαν και ποιοι όχι 55 ηλεκτρονικά ψήφισαν οι πάντας πέρας υιοθετείται με μία ψήφο μόνο 13 με προφορική προπολογία και απαιτεί ε, απαιτείται χωριτηματική ψηφοφορία όχι ωραία προφορική ως υπέρ της προφορικής κατά αποχές υιοθετείται και τώρα ερχόμαστε στο πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται Τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τέσσερο τέταρτο υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τέντα είναι ταυτόσιμο. Θεματική ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, υιοθετείται τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται επίσης συμβαστική πρόταση δέλτα δε υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 59 σε τέσσερα μέρη το 59 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε το δεύτερο μέρος παρακαλώ με τις κάρτες σας. Ψήφισαν οι πάντες, πέρας. Υιοθετείται το δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές Απερίφθητο το μέρος, τέταρτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 16 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε το 16 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψήψαν οι πάντες, πέρας, Απερίφθη. Απερίφθη. Θεματική. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Καταπίφθη το δεύτερο μέρος. 17 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 19 υπέρ κατά απερίφθη το προηγείο 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 20 υπέρ κατά αποχές το 21 συγγνώμη ξανά το 21 ξανά το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Υιοθετείται 21 με 18. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε το 23. Λοιπόν, οι πάντες πέρας καταπίπτει 21-21 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 24 υπέρ μια στιγμή καταπίπτει 24-25 με τη ψηφοφορία σε τρία μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απερίφθη Αφού φεύγει το πρώτο, έχει νόημα να ψηφίσουν τα υπόλοιπα. Ο Στο τρίτο μέρος, μα. Γιατί το δεύτερο καταπίπτει. Το δεύτερο πέφτει. Πάμε στο τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθηκε το τρίτο μέρος. 26 τροπολογία υπέρ. Τρόπο κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 27 υπέρ κατά υιοθετείται 3 υπέρ κατά χες υιοθετείται 29, δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 30 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 31 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 32 υπέρ, κατά αποχές απεριφθεί. 33 σε δύο μέρη Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Δεύτερο μέρος, καταπίπτει το δεύτερο μέρος. 34 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 35 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 4 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 37 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 28 καταπίπτει 39 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. το 40 σε δύο μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 41 είναι ταυτόσιμο υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 42 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 44 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως υιοθετείτε και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ για το τελικό κείμενο έτσι όπως τροποποιήθηκε ψήφισαν οι πάντες πέρας 42 υπέρ ομοφωνία ουδής κατά Ουδεμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή παρακαλώ. Μάρτιν, ζήτησε το λόγο παρακαλώ. Ο Χάντς Πέτερ Μάρτιν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία ε, αντικειμενική και η γραμματεία σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άψογα όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ραντεβού το απόγευμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον